I would like to welcome you to this... Να σας καλυσ... καλωσορίσω και να σας καλημερίσω. Παρακαλώ να καθίσουμε όλοι για να ξεκινήσουμε τις συνεδρίασή μας. So my first item is the, the, uh, the uh, adoption. Πρώτο θέμα. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξη εγκρίνεται. Έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής τα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει και ενστάσει μπορούμε να τα εγκρίνουμε, τα πρακτικά δηλαδή τη συνεδρίασης τη 26 Φεβρουαρίου. Να κάνω κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά μου. Καλωσορίζουμε νέα administrator, την Z. Καλώς ήρθατε. Και σας παρακαλώ να είστε καλοί μαζί της. Η Κλέρ έχει δουλέψει, ε, είναι από τη Γαλλία και έχει ε, δουλέψει στην ε, Επιτροπή ΕΝΒΗ και στο Τμήμα Πολιτικής. Επίσης, η ακρόαση για το δικαίωμα στην υποβολή αιτήσεων θα γίνει 23 Ιουνίου το πρωί. Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας θα γίνει 4 και 5 Μαΐου και θα έχουμε εκπροσώπους και από την Επιτροπή Αναφορών του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Θα έρθει επίσης ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς στις 5 Μαΐου στις 3 το απόγευμα. Ελπίζω να προσέλθετε μαζικά σε αυτές τις δύο πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις. Όσον αφορά την συνάντηση με τον κύριο Τίμερμανς, ε, θα πρότεινα πρώτα να δώσουμε το λόγο στους συντονιστές και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία Catch the Eye. Συμφωνείτε? Ωραία. Δεν υπάρχουν θέματα στα διάφορα. Περνάω λοιπόν στις αποφάσεις των συντονιστών που λάβαμε στη συνεδρία των Τενστών μόλις πριν από λίγο. Έγκριση της ε, ημέρας διάταξης του Μαΐου. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές σύμφωνα με τις ε, συζητήσεις που είχαμε και θα αποσταλεί σε σας για γραπτή έγκριση. Και οι ισπανικές αναφορές θα αναβληθούν για την συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου λόγω του ότι διεξάγονται εκλογές στη χώρα. Υπάρχει ένα θέμα από τους σοσιαλιστές για την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όσον αφορά την κατάσταση στην ε, Μεσόγειο και μια ολιστική προσέγγιση προς το ζήτημα της ε, μετανάστευσης. Υπάρχει προθεσμία 23 Απριλίου για ενστάσεις όσον αφορά τον κατεξοδότηση κανονισμό ε, σχετικά με τον κανονισμό ECI για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Οι συστάσεις έγιναν αποδεκτές όπως τις πρότεινα εγώ με εξαίρεση το 1062 του 14 αναφορά που κηρύχθηκε μη παραδεκτή θα, υπάρχουν, ε, θα δοθούν δύο επιπλέον μήνες στους αναφέροντες, στον αναφέροντα για να υποβάλει νέες πληροφορίες. Και ε, έχουμε συζητήσει πολλά θέματα στους συντονιστές, θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω όλα. Για τις διερευνητικές επισκέψεις. για τις διερευνητικές επισκέψεις. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία στο τέλος της φετινής χρονιάς λόγω του, γεγονός ότι, του γεγονότος ότι είχαμε ε, μπαλιάζ και συμπεριλαμβάνεται και η Ισπανία. Θα συμφωνήσουν οι συντονιστές μεταξύ τους για το πού θα πάμε και για το 2016 ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες να επισκεφθούμε τους πολίτες εκεί που ζουν. Ελπίζουμε δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε τρεις ίσως και κάποιες παραπάνω διερευνητικές επισκέψεις και αυτό αντικατοπτρίζει και την θέση και την επιθυμία όλων των πολιτών να επανέλθουμε στους πολίτες και να προσπαθήσουμε να γεφερώσουμε αυτό το κενό που αισθάνονται πολλοί πολίτες ότι υπάρχει μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ιδίων υπήρχε ένα αίτημα για επανέρεξη συζήτησης για την αναφορά, για συγκεκριμένη αναφορά από την κυρία Βαλέντσα. Αποφασίσαμε να το συζητήσουμε στο πλαίσιο των νέων κατευθυντηρίων γραμμών της ΠΕΤΗ που θα συζητηθεί στο, στην επόμενη συνεδρίαση συντονιστών. Επίσης υπήρχε θέμα από το EFDD και την κυρία Εύη να ξανανοίξει τη συζήτηση για το Jugendamt το οποίο επίσης θα συζητηθεί ε, με την ευκαιρία της επίσκεψης των ε, ε, συναδέλφων από τον Bundestag. Υπήρξε ένα αίτημα από τους Πρασίνους για να ξανανοίξει συζήτηση για τη 1503 του 13 και αποφασίστηκε να μην ξανανοίξει συζήτηση. Σχόλια για την διαδικτυακή πύλη ΠΕΤΗ. Η Γραμματεία θα εξετάσει αυτά που ακούστηκαν και θα επανέλθει δίνοντας περισσότερες πληροφορίες στα επόμενα βήματα καθώς θα υλοποιείται το έργο αυτό. Υπάρχει και η ε, επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ουαλίας, η οποία θα μας επισκεφτεί τον ε, ε, Ιούνιο και θα παρακολουθήσει και την ακρόαση δικαίωμα στην υποβολή αναφορών, που θεωρούμε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον και ε, ως συντονιστές ε, προτείνουμε να διοργανώνεται κάθε χρόνο συνάντηση με τις Επιτροπές Αναφορών των Εθνικών Κοινοβουλίων για την ανταλλαγή βέλτιστων προεκτικών. Ε, και αυτή η πρόταση εγκρίθηκε από τους συντονιστές. Υπήρχε και η, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που απέτυχε σχετικά με τον ορισμό ορίου ταχύτητας 30 ε, χιλιόμετρων την ώρα. αποφασίσαμε να μην αναλάβουμε καμία δράση όπως έχουμε δικαίωμα για, ε, αποφασίστηκε επίσης να ζητήσουμε από, την, από το Τμήμα Πολιτικής να εκπονήσει μελέτη για την υιοθεσία χωρίς συγκατάθεση, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει διερευνηθεί. Αυτά. Είχαμε μια πολύ γόνιμη και έντονη, θα έλεγα, συζήτηση στους συντονιστές. Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο θέμα 7 ψηφοφορία σχετικά με τη γνωμοδότηση, σχετικά με τι συστάσεις προ την Επιτροπή όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. TTIP. Ελπίζω να έχετε μαζί σα τι κάρτε σα, Παρακαλώ βάλτε, τα στα, στα μηχανηματάκια. Ο λόγο στη Μάργκρετ. Το είπα και στου συντονιστέ. Νομίζω ότι η ψηφοφορία Α, η γνωμοδότηση αυτή ε, έχει τύχει απαράδεκτης μεταχείρισης. Τροπολογίες από τις ε, ομάδες ε, έχουν αγνοηθεί με ευθύνη του μεγάλου συνεσπισμού και ακόμη και αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ειδική ψηφοφορία, συγγνώμη που κάνω μια τέτοια πολιτική τοποθέτηση, συνήθως όταν δεν συμφωνείς με κάποια συμβαστική πρόταση, Μπορεί να υποβάλει μια δική σου τροπολογία αν δεν, είναι, αν δεν έρχεται σε αντίθεση ή αν δεν καλύπτεται ήδη. Αν είναι συμπληρωματική η τροπολογία θα πρέπει να τεθεί στην ψηφοφορία. Φυσικά μπορεί να καταψηφιστεί, αλλά το να αγνοείται μια τροπολογία που έχει ε, προταθεί είναι νομίζω μια διαδικασία, μια ε, συμπεριφορά παράδεκτη η 101 θα πρέπει τουλάχιστον να ψηφιστεί και θα πρέπει να διασφαλίσουμε στο μέλλον ότι οι τροπολογίε που δεν καλύπτονται από, άλλες, από την συμβαστική πρόταση και δεν έρχονται σε αντίθεση μαζί τη θα πρέπει να προστίθενται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ε, μιλάω για την τροπολογία 101 ε, σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ε, κάποιες χημικές ουσίες, ότι θα πρέπει να εξαιρούνται από το TTIP. Εγώ, λέει η Πρόεδρος, έχω το δικαίωμα να αποφασίσω τι τίθεται στην πληροφορία στην Επιτροπή. Έχετε βεβαίως δικαίωμα να υποβάλλετε τροπολογίες και να, ζητείτε να, να ζητάτε να γίνεται ξεχωριστή ψηφοφορία. Ωραία. Επί της διαδικασίας. Η κυρία Κέρτεν Ντόλεν. Εκ μέρους των σοσιαλιστών. Υπάρχει στον κατάλογο ψηφοφορίας μια προφορική τροπολογία για το 12 και θα ήθελα να πω εκ μέρους των σοσιαλιστών ότι εμείς διαφωνούμε με αυτήν την ε, προφορική τροπολογία. This κυρία Αλπιόλη έχει ζητήσει το λόγο. Σύντομα, σύντομα. Συμφωνούμε με αυτό που ακούσαμε. Και στην περίπτωσή μας ε, της αριστεράς ε, είχαμε, δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία. Θέλουμε όμως να ψηφιστούν γιατί είναι συμπληρωματικές. Ε, ε μερικές φορές στις συμβαστικές τροπολογίες αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που είχαμε πει ναι εμείς στις επιμέρους Ξεχωριστή ψηφοφορία ζητάτε. Εντάξει, θα γίνει. Can I now proceed to the... Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία, ε, γνωμοδότηση Βαλέσσα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Α, ζητώ συγγνώμη, τμήματική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 για το πρώτο τμήμα με την προφορική τροπολογία. Όχι, σας ζητώ συγγνώμη, η προφορική τροπολογία απερίφθη. Επομένω ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Μάλλον ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο εδώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Έναρξη ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έχει δύο επιπλέον. Δύο παραπάνω. Δύο περισσεύουν. Δηλαδή... Εντάξει, διορθώθηκε. Διορθώθηκε, λέει η πρόεδρο. Εντάξει, κλείνει επέρ ψηφοφορία. Και με 11 ψήφου υπέρ 15 κατά απορρίπτεται. για το δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορία. Θα το κάνουμε και αυτό ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Έναρξη ψηφοφορία. Για το δεύτερο, ναι, για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε τώρα. είναι για το δεύτερο τμήμα και έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα είναι ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Με 18 ψήφους υπέρ και 12 κατά εγκρίνεται. Προλογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αυτό πρέπει να το ελέγξουμε νομίζω. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά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 Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Και πάλι ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη ψηφοφορίας. Ε, ε, συγγνώμη, ε, ακόμα μπορείτε να ψηφίσετε. Αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 24 για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ας το ελέγξουμε έναρξη ψηφοφορίας πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε. Γιατί όλα αλλάζεται. Άποψη μάλλον εννοεί η Πρόεδρος. Επομένω, το κάνουμε σωστά. Να είμαστε σίγουροι. Έναρξη ψηφοφορίας. θα με βοηθούσε αν οι συντονιστέ των πολιτικών ομάδων δείχνουν την άποψη της θέσης, του κόμματο του. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 ε, υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, 35 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε Όλα αλλάζεται, όλα αλλάζεται. Δεν υπάρχει καμία συνοχή στον τρόπο που ψηφίζουν οι ομάδες. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 36, 36 τριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 42 υπέρ. Ζητήσατε να ελέγξουμε για τις 41. 41 έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Είδατε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται λέει η πρόεδρος. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε όμως για τη 44 ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξης. Πέρας ψηφοφορία. Κοίτα εδώ. 22 κατά. Ναι, αλλά θα με βοηθούσε οι συντονιστέ των πολιτικών ομάδων να μου δείχνουν να ψηφίζουν. 45 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται, 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 47 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται, ωραία, να ελέγξουμε, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφορίας, Πέρας και και εγκρίνεται. 48. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, μη λέτε όχι, παρακαλώ ζητάτε έλεγχο. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία. 54. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πενήντα έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μη λέτε σας παρακαλώ όχι να ζητάτε έλεγχο. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία για, για την τροπολογία 56. Πέραση ψηφοφορία για την τροπολογία 56. Και εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε στη βασική πρόταση. Τροπολογία, με συγχωρείτε, 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας για την τροπολογία 58.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 κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά όμως εντάξει ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε για την τροπολογία 67 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Πρώτο, ε, τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86 όχι, συγγνώμη, περιμένετε. Υπάρχει και άλλη συμβαστική τροπολογία. Η συμβαστική τροπολογία 4, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζητήθηκε από τους πρασίνους να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 101. Ωραία. Υπέρ της τροπολογίας 101. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κάθε φορά που κάποιος συνάδελφος ε, ζητά ηλεκτρονική ψηφοφορία, την κάνουμε. 105, 104, ε, με συγχωρείτε, τροπολογία 104, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 7, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας για, το, για την τροπολογία 107. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και στο δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, ωραία. Βεβαίως, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αφού θέλετε. Κανένα πρόβλημα. Ένας προφορίας. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Εκατόν δεκατέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίση. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται και αυτή. Να ψηφίσουμε τώρα για, την, για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό της και θα το κάνουμε αυτό ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. χρειαζόμαστε λίγες ακόμα ψήφους. Πρέπει άλλος ένας να ψηφίσει. Αν δεν ψηφίσει, θα τελειώσει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία.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 Έχει αποσεχθεί. Συμβαστική πρόταση, τροπολογία, με συγχωρείτε, 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 έχει αποσυρθεί και πάμε στην συμβαστική τροπολογία. Ε, με συγχωρείτε, 2, 2. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 έχει αποσυρθεί 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, εντάξει, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, ένα ψηφοφορίας. Ψηφοφορία για την τροπολογία 23. Ηλεκτρονικά. και να ξαναζητήσω από τους συντονιστές να υποδεικνύουν τι ψηφίζουν οι ομάδες τους. Είμαι κι εγώ μέλος, ξέρετε. Πρέπει κι εγώ να ξέρω τι θα ψηφίσω. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, με συγχωρείτε, εγκρίνεται. Ναι, ε, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 έχει αποσυρθεί 50 υπέρ κατά εγκρίνεται 55 υπέρ 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 50, συγγνώμη, 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ α καταπίπτει 66 67, συγγνώμη. Ναι, έχουμε ψηφίσει ήδη. Okay, the request by the Greens is... Έτοιμα των Πρασίνων είναι η τροπολογία 66 να τεθεί σε ψηφοφορία με το συμπληρωματικό τμήμα που δεν συμπεριλαμβανόταν. Οπότε το, βάζω σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ του συμπληρωματικού τμήματος που θεωρούν οι πράσινοι ότι δεν καλύπτεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Για την τροπολογία 66. Έναρξη ψηφοφορίας. And I close it. ψηφοφορίας. rejected. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 72 έναρξη ψηφοφορίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ψηφίστε παρακαλώ τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 έχει αποσυρθεί 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92. Η Σολεδάδη, η συγκίτρια ζητά το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αδούδα. Ε, μια αμφιβολία τρέφω. Η 82 έχει καταπέσει από τη στιγμή που η 55 εγκρίνεται. Η 55 εγκρίθηκε. Γιατί λοιπόν να ψηφίσουμε και την 82 τώρα. Καταπίπτει από τη στιγμή που έχει υπερψηφιστεί 55. Ναι, το, το, το ελέγξαμε, έχετε απόλυτα δίκιο, ναι. Εντάξει, άρα λοιπόν την αφαιρούμε από τον κατάλογο ψηφοφορίας. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1.96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ζήτησε κάποιος να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 96. Ναι, βεβαίως. 96 λοιπόν, έναρξη ψηφοφορίας. πέρα στις ψηφοφορίας. Και πράγματι εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε για την 97 έναρξη 97 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μικρή, με, ένα, με μία ψήφο διαφορά. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ψηφοφορίας. η ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια, Σολεδάδ. Σας ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία μας πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Χρειάζεται να προχωρήσουμε στη συζήτηση των διαφόρων αναφορών και ξεκινούμε την αφορά 9, ε, σημείο 9 της σημερινής διάταξης, Πολ Στέφαν, αυστριακής κατηγορής, για τον οικότοπο Μάτι Χαλ. Ο αριθμός είναι 1004 του 2014. Καλωσορίζω τον αναφέροντα, τον κύριο Πολ Στέφαν, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μας ε, κάνει την παρουσίασή του με τη χρήση ενός PowerPoint και μετά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε γιατί μας πήρε τόσο πολύ χρόνο η ψηφοφορία, αλλά αυτό που συνήθως κάνουμε στην Επιτροπή είναι να συζητάμε τις αναφορές. Έχετε το λόγο για 4-5 λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας χαιρετήσω, να σας συστηθώ. Είμαι ο Πάουλ Στέφαν, είμαι πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου που είναι και αναγνωσμένο από το Υπουργείο μας ε, Κότοπος Μάτικτε. Αντικείμενο της καταγγελίας μας είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος Β147 μεταξύ Μπράουνα Οαμίν και Σράλς Βάλχεν. Ο σχεδιασμός του συνολικού έργου έχει ολοκληρωθεί και θα αποτελέσει νέο δρόμο παράλληλα προς την ε, υπάρχουσα, αυτό στον υπάρχοντα ε, κινητόδρομο Β 147. Το έργο αυτό έχει από τους αρμόδιους πολιτικούς χωριστεί σε πέντε τμήματα. Και έτσι αιτιολογείται ότι δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τον ε, νόμο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 2000. Το πρώτο τμήμα θα είναι το Μάτι Χόφεν Μούντερφινγκ ε, ε, μεγέθους 9 χιλιόμετρων. Στο πνεύμα της συνομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν επιτρέπεται η κατάτμιση των έργων και δεν μπορεί να παρακαμφθούν οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία περιεκτήμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, μέσω της ε, κατάτμισης των έργων. Κάτι αντίστοιχο ε, έχει συμβεί με, την, με τον αυτοκινητόδρομο Α94. Υπάρχει δηλαδή, κατασκευάζεται ένας αυτοκινητόδρομος που περνά μέσα από πυκνά κατοικημένη περιοχή. Επίσης, ε, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συνολικού έργου θα είναι υψηλότερες αθρηστικά από τον, των επεμέρους τμήματων του έργου. Όλος ο νέος αυτοκινητόδρομος Β147 θα έχει μήκος 40 χιλιόμετρα. Το Σάλχεν για παράδειγμα η κομμόπολη αυτή θα ε, διχοτομηθεί από αυτόν τον ε, αυτοκινητόδρομο. Το βλέπετε και εδώ στο χάρτη. Στη βάση των ε, στοιχείων που υπάρχουν τίθεται κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων και των επόμενων γενεών. Και η μη εκπόνηση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιτεώσεων βασίζεται σε μια τακτική σαλαμοποίησης ενώ οι περιβαλλοντικέ επιπτώσει οξύνονται ακόμη περισσότερο μέσω της μερικής ε, επέκτασης. Εμείς θεωρούμε και ζητούμε το τμήμα από Μπράουνάου μέχρι το Στρας Βάλχεν να ελεγχθεί και να εκπονηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων γι' αυτό, όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο. Εμείς ως σύλλογος δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα με βάση τη διαδικασία που προβλέπετε να κάνουμε τίποτα. Επίσης δεν μας δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, σύμφωνα με την Σύμβαση Άρχους, προβλέπεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε δικαστική προστασία σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Αλλά είναι ένα δικαίωμα το οποίο εμείς δεν έχουμε την ε, δυνατότητα να το ασκήσουμε. Ακριβώς γιατί δεν ε, μας δίνεται πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπτώσεις του έργου για μας είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού θα αυξηθούν δραματικά. 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα καλλιεργήσιμης γης θα καταστραφούν. Το Σάλχεν, ένα χωριό με 3.500 κατοίκους, θα διχοτομηθεί, ενώ επίσης αυξάνεται ο κίνδυνο πλημμυρών στην κοιλάδα από την οποία θα περνάει ο αυτοκινητόδρομος. Επίσης, η χρησιμότητα του έργου αυτού είναι απόλυτα δυσανάλογη με το υψηλότατο κόστος του έργου αυτού. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική μελέτη του καθηγητή Μακούν του Πολυτεχνείου της Βιέννης που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015. Η παράκληση μας σε εσά είναι ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί επίγουσα διαδικασία. Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα και εμεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τίποτα. Παρακαλούμε να καλέσετε την Αυστριακή Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αλλά και την τοπική κυβέρνηση της Άνω Αυστρίας να επιβάλλει την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλο το έργο όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο του 2000. Βοηθήστε μας ώστε η Αυστρία να θέσει στη διάθεσή μας αυτά που προβλέπονται στην Σύμβαση Άρχους. Επίσης, θα μπορούσατε ίσως να ε, καλέσετε την κυβέρνηση και την, ε, τις περιφερειακές αρχές να προχωρήσουν σε ε, μια μελέτη για την κατασκευή διατροπικών μεταφορών. Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να μην μας λαμβάνουν υπόψη σοβαρά μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αλλά και στην Αυστρία. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι πολιτικοί προσπαθούν να παρακάμψουν ισχύοντα νόμο και αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει, υπάρχουν, υπάρχουν αδυναμίες ως προς τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επίσης, να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι υπάρχετε και σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι επιτέλους μας κάνετε και αισθανόμαστε ότι είμαστε σημαντική. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που μας δώσατε στο θέμα μας και σας εύχομαι ε, μια γόνιμη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στέφαν για το γεγονός ότι ταξιδέψατε μέχρι εδώ στις Βρυξέλλες και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, τον κύριο Μάρκ Όλβερ Χάιτκαμ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, ε, ευχαριστώ και τον αναφέροντα για τις για τα στοιχεία του. Θα ήθελα να σας πω ότι πρώτον έχουμε λάβει την αναφορά μόλις χθες, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να τοποθετηθώ ε, οριστικά επί του θέματος. Φαίνεται ότι από μια πρώτη μελέτη και εξέταση των ε, ε, εγγράφων φαίνεται ότι πράγματι είναι αιτιολογημένη η αναφορά αυτή και θα πρέπει να την ε, εξετάσουμε ε, ως προς τις λεπτομέρειές της. Ο αναφέρον έθεσε προς δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αυτή η, τακτική της αλαμοποίησης, όπως ε, λέει και ο ίδιος. Συμφωνούμε ως Κομισιόν ότι με βάση την ομολογία του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ισχύει όταν ένα συνολικό σχέδιο επίτηδες κατανέμεται και χωρίζεται σε τμήματα για να παρακαμφθεί η υποχρέωση εκπόνησης ε, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν επιτρέπεται. Να συνοψίσω λοιπόν ποια είναι η δική μας αντίληψη. Ο Αυστριακός νόμος προβλέπει ε, όριο 10 χιλιόμετρων, μήκο 10 χιλιόμετρων για την ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα πρέπει να ε, ελέγχονται και αθρηστικά, σορευτικά οι επιπτώσεις όταν ε, κατασκευάζεται ένα τέτοιο είδους έργο. Ο αναφέρον ανέφερε ότι ο συνολικός σχεδιασμός του έργου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ε, εμείς ε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε, ε, ισχύει αυτό, πώς, πώς, πώς, πώς τεκμηριώνεται αυτό με βάση τις εγκρίσεις. Εμείς αυτό που, βλέπουμε είναι ότι έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής τρία ε, υποέργα να το πω έτσι, εκ των οποίων το πρώτο έχει εγκριθεί, το δεύτερο βρίσκεται στη διαδικασία της έγκρισης, ενώ το τρίτο δεν έχει καν μπει στη διαδικασία της ε, αδειοδότησης, ε, της έγκρισης. Επίσης, μια παρατήρηση να κάνω. Όταν κάποιο δεύτερο έργο, σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κάποιο δεύτερο έργο στον ίδιο χώρο, θα πρέπει και σωρευτικά σε αυτή την περίπτωση να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε, συνδυασμό δηλαδή με το πρώτο έργο. Η Κομισιόν, όπως είπα και αρχικά, ε, θα ελέγξει τα στοιχεία και θα τοποθετηθεί γραπτά το δεύτερο θέμα που έθεσε προς συζήτηση ο αναφέρον είναι αυτή η, κατηγορία ότι δεν ε, εφαρμόζεται πλήρως η σύμβαση άρχους. Είπε ότι είναι πρόεδρος ενός αναγνωρισμένου από το Υπουργείο και τον νόμο ε, Αυστριακού Περιβαλλοντικού Συλλόγου. Θεωρούμε ότι με αυτήν την ιδιότητα δεν μπορεί να ζητήσει ε, μια διαδικασία διαπίστωσης. Θα μπορούσε ε, ο Σύλλογος να προσφύγει στα δικαστήρια για την εφαρμογή της Σύμβασης Άρχους και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ε, απόφαση αρνητική έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στα δικαστήρια. Να σας πω από τώρα, αλλά επιφυλασσόμενος της ε, ε, περαιτέρω εξέτασης που θα κάνει η Κομισιόν, ε, ενδέχεται λοιπόν να υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει τελικά αρνητική απόφαση την οποία θα μπορούσατε να καταγγείλετε θα μπορούσατε να προσφύγετε στα δικαστήρια για το γεγονός ότι δεν έχετε την, ε, το δικαίωμα να ζητήσετε δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή εκδικάζεται και μια παρόμοια υπόθεση κατά της Αυστρίας Σύντομα λοιπόν, δεν, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε, αλλά σύντομα αναμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ελπίζουμε να τοποθετείτε και ως προς το θέμα της πρόσβασης των περιβαλλοντικών συλλόγων σε δικαστική προσφυγή θα το αναλύσουμε εμείς και μόλις έχουμε ε, πληροφορίες βεβαίως θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα, σας θέσουμε, θα θέσουμε και στη δική σας διάθεση τις πληροφορίες αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αναφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στους συναδέλφους, ο κύριος Μπέκερ. Παρακαλώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Αν δεν είναι απαραίτητο να πάρετε το λόγο, παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει μισή ώρα. Κύριε, κύριε Μπέκερ, έχετε δύο λεπτά για να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ εκπρόσωπε της Κομισιόν, αγαπητέ αναφέροντα. Να πω καταρχάς ότι έχουμε με μια ε, επίγουσα κατάσταση, έχουμε κάνει μια γιατί το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός των επόμενων εβδομάδων και θα ήθελα να ε, ε, πω ότι δεν καταλαβαίνω πώς ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αναφέρει ότι μόλις χθες έλαβε τα έγγραφα. Πρέπει να εξηγήσει τι εννοεί. Κατά τα άλλα, είναι σαφές ότι η σοβαρότατη καταγγελία των αναφερόντων περί παράκαμψης της νομοθεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να ελεγχθεί από την Κομισιόν και ε, ευχαριστώ για το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν προφασίστηκε την ε, αργή, την ε, χθεσινή μόλις παραλαβή των εγγράφων και για το γεγονός ότι τοποθετήθηκε επί της ουσίας. Ακριβώς λοιπόν επειδή επίκειται η έναρξη των εργασιών θα πρέπει να αναλυθούν γρήγορα πρωτοβουλίες και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ε, ικανοποιηθεί όλες οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να αναλυθούν οι κατάλληλες ε, δράσεις. Είναι σοβαρότατο θέμα αν μια αρχή προσπαθεί να παρακάμψει την ισχύουσα νομοθεσία, γι' αυτό θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ε, καλέσουμε να τοποθετηθεί και η Αυστρία. Ο Πέτερ Γιάρ. Ναι, συμφωνώ. Έχουμε μάλλον ε, ένα θέμα εδώ που αφορά ιδιαίτερα την Αυστρία. Είχαμε ένα παρόμοια, παρόμοιο θέμα πρόσφατα ε, όπου δεν είχε εκπονηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ θα έπρεπε κανονικά να είχε εκπονηθεί. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξή. Η Κομισιόν διαπίστωσε σωστά. Για τα πρώτα 10 χιλιόμετρα δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Αν υπάρξει διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν επεκτάσεις, δεν θα υπάρξουν άλλες κατασκευές έργων. Αν όμως κάποιος θέλει στη συνέχεια να επεκτείνει το έργο είναι σαφές. Δεν έχει νόημα στη δεύτερη φάση να απαγορεύσουμε την, ε, την εκτέλεση των έργων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τώρα πληροφορίες από την Αυστρία να μας πει η Αυστρία ποια ακριβώς είναι τα σχέδιά της για το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να ζητά το λόγο. Να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και να ζητήσουμε από τις αυστριακές αρχές να μας παράσχουν πληροφορίες. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Και για, ο ταχύτερος τρόπος για να λάβουμε τις πληροφορίες αυτές είναι να επικοινωνήσουμε με την μόνιμη αντιπροσωπεία της Αυστρίας εδώ στις Βρυξέλλες και να, ε, να συνεχίσει η διαδικασία από εκεί. Κύριε Αναφέροντα, είστε ικανοποιημένος με αυτή την πρόταση. Αν είστε εσείς είμαι και εγώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε... Όχι. Έχω εδώ για την Κομισιόν έναν χάρτη όπου αποδεικνύεται ότι το έργο αυτό ε, θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί. Ε, ε, έχει ήδη δηλαδή σχεδιαστεί. Ε, να σας πω μάλιστα ότι το έργο αυτό στο σύνολό του μπορούσε κανείς να το βρει στην σχετική ιστοσελίδα μέχρι το 2010, τώρα πια όχι. Ωραία, σας συνιστώ λοιπόν να συζητήσετε με την Κομισιόν. Εμείς θα επικοινωνήσουμε από την πλευρά μας με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Αυστρίας εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι επιστροφής και Τώρα, η επόμενη αναφορά που θα συζητήσουμε είναι η 1833 του 2013 της Γκίζελα Urban και της Γκαμπριέλ Μέντσνερ εκ μέρους ε, συλλόγων για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων. Στρέφομαι προς εσάς. Ελπίζω να είστε εδώ. Πού, είναι οι αναφέροντες, οι αναφέρουσες. Α, εδώ είστε. Παρακαλώ καθίστε και δίνω το λόγο σε εσά. Έχετε πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Could we get started as soon as possible? Να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό. Έχετε και, και βιντεάκι να μας δείξετε, οπότε Παρακαλώ, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Αγαπητοί Πρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών, αγαπητοί ε, βουλευτές, τον Οκτώβριο του 2013 υποβάλαμε αναφορά με τίτλο «Σταματήστε το ρίτς, καταργήστε τα πειράματα στα ζώα». 1η Απριλίου 2014 η Επιτροπή Αναφορών κήρυξε την, την αναφορά μας ως παραδεκτή. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε και μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο αμέτρητα ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους. Ε, πιστεύουμε ότι τα πειράματα σε ζώα είναι ηθικά αναξιόπιστα και επιστημονικά επίσης. Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς την ε, χρήση ζώων όπως αυτές που έχουν προτείνει ο κύριος ε, ο Δόκτωρ Κλόντ και Άντρε Μάχε. Δυστυχώς όμως αυτές οι εναλλακτικέ μέθοδοι δεν έχουν επαληθευτεί. Αλλά κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι ούτε τα πειράματα στα ζώα έχουν ποτέ επαληθευτεί ως προς την αξιοπιστία τους. Κάθε 10 δευτερόλεπτα μόνο στη Γερμανία πεθαίνει ένα ζώο στο πλαίσιο πειράματος σε ζώα. Στην ε, Γερμανία κάθε χρόνο είναι 3 εκατομμύρια τα ζώα που χάνουν τη ζωή τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12 εκατομμύρια. Ενώ περίπου 58.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στη Γερμανία από παρενέργειες φαρμάκων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Και μάλιστα είναι ο, η αιτία θανάτου υπαριθμών 4. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει επιστημονική κατάρρηση ώστε να υποψιαστεί ότι τα απορίσματα που ε, βγαίνουν από ε, πειράματα σε ζώα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο είδος του, κάθε, του εκάστοτε ζώου. Για, για να μην πω μάλιστα ότι τα πορίσματα αφορούν το εκάστοτε ζώο στο οποίο διενεργήθηκε το πείραμα. Με βάση την, την κοινή λογική μπορεί κανείς να καταλάβει ότι αποτελέσματα πειραμάτων που έχουν διεξαχθεί σε αρουραίους δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι αυτόματα και ευθύγραμμα σε ανθρώπους. Θα θέλαμε να σας, δώσουμε, να σας δείξουμε ένα βιντεάκι και να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι ευρωπαϊκοί νόμοι αλλά και εθνικές διατάξεις προβλέπουν ότι πολλές φορές θα πρέπει να γίνονται δοκιμές και σε μη τροκτικά, εκτός από τα τροκτικά και σε, ζώα που δεν είναι τροκτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για σκύλους και γίνονται πειράματα ε, για τον έλεγχο παρασιτοκτόνων και φυτοφαρμάκων. Εδώ μιλάμε, στο συγκεκριμένο βιντεάκι θα δείτε ε, την περίπτωση της ε, χημικής ουσίας τριμεθυλοφοσφίνης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 Προφανώς υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε μελετήσει την αναφορά σας. Η Επιτροπή μας έχει ενημερωθεί για όλες τις προφορίες που μας έχετε παράσχει, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ε, προχωρήσουμε. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε και στη συνέχεια θα δώσω τον ε, λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ωραία, αφού δεν είδαμε το βιντεάκι θα σας το περιγράψω. Ε, μιλάμε για ένα ε, εργαστήριο στην Ελβετία και μια μελέτη για ε, φυτοφάρμακο παραστοκτόνο το, την, τον τριμεθυλοφοσφαίνη. Και εκεί σε αυτό το βίντεο αποδεικνύεται η απίστευτη, η αδιανόητη βία που, υφίστανται, τα ζώα αυτά. Εμφανίζονται επιστήμονες να χώνουν το χέρι τους με, γάντι μέσα στο στόμα των ζώων. Υπάρχουν, είναι απίστευτα τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονται ε, τα ζώα αυτά. Την εκατοστή Πέντη η μέρα πεθαίνει και το τελευταίο ζώο. Με ποιο δικαίωμα υποβλήθηκαν τα ζωάκια αυτά σε αυτά τα βασανιστήρια. Δεν είναι ανήθικο το να δηλητηριάζεις πλάσματα, ζώντα, όντα. Από μελέτη στις ε, διατάξεις ελέγχου του ΡΙΤΣ, της οδηγίας για τα βιοκτώνα και της οδηγίας για τα ε, παρασιτοκτώνα αλλά και της οδηγίας για τα νέα τρόφιμα απέδειξε ότι πολλές φορές οι απαιτήσει που προβλέπονται στην νομοθεσία δεν ανταποκρίνονται στο τρέχον επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Συγγνώμη, ο προηγούμενος αναφέρον είχε και αυτός λίγο παραπάνω χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει η Πρόεδρος, το θέμα. Ε, την έχουμε μελετήσει. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το βίντεο. Μπορούμε να δώσουμε τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και στη συνέχεια στους συναδέλφους. Και μετά μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση. Συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία, ε? Οπότε δίνω το λόγο στον Κάρη Κίλιαν από την Κομισιόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό περιθώριο που μου δίνετε, γιατί έχουμε ήδη δώσει απαντήσεις κατά το παρελθόν, δηλαδή στην πρώτη ακρόαση που έχει γίνει για την πρώτη αναφορά. Θα σταθώ σε λίγα κεντρικά ζητήματα που φύγει αυτή η αναφορά. Που εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το ποια είναι η αξία η επιστημονική να χρησιμοποιούνται τέτοια ε, πειραματόζωα, κατά πόσον είναι διαθέσιμα αυτά τα πειραματόζωα για το, την τοξικολογία και τρίτον, ποιε είναι οι απαιτήσει τη ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα του κανονικού, ε, κανονισμού REACH. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα κατηγορηματικά να πω ότι αντιτιθέμεθα σε αυτή τη θέση την οποία εκφράστηκε και στην ε, αναφορά αλλά και κατά τον λόγο σας τώρα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ένα ζώο ως μοντέλο επιστημονικό για να μελετηθούν οι άνθρωποι. Αυτό δεν ισχύει τα τελευταίου, τους τελευταίους αιώνες έχουμε καταφέρει, τα τελευταία 100 ε, χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε πρόοδο στην ιατρική ε, εξετάζοντας φάρμακα και ουσίες πρώτα απ' όλα σε ζώα, σε πειραματόζα ζώα το οποίο αποδεικνύει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πειραματόζωα ως μοντέλο για την ανθρώπινη ύπαρξη, για τους ανθρώπους. Έχει όρια βέβαια η επιστημονική γνώση και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα αντιληφθούμε αυτά και να τα αναγνωρίσουμε. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα και αυτές Μα έχουν δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πολύ καλύτερα πώ λειτουργούν οι μοριακοί μηχανισμοί στο κύτταρο και αυτή η μοριακή βιολογία πλέον χρησιμοποιείται και για να συμπληρώνει αλλά και ορισμένε φορές να αντικαθιστά τα πειράματα σε ζώα. για να επιβεβαιώνει με μεγαλύτερη ασφάλεια τα αποτελέσματα πιθανώς που έχουν ε, αντιληφθεί από ε, πειράματα σε ζώα. Ωστόσο, αυτή η επιπλέον γνώση που αποκτάμε είναι απλώς κάποια κομμάτια του παζλ δεν έχουμε στη διάθεσή μας ένα πλήρες μοντέλο για το τι συμβαίνει στο επίπεδο των πολυκύτταρων οργανισμών. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε τα, ακόμα τα πειράματα σε ζώα. Και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ανάγκη και για το προβλέψιμο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για την ιατρική. Αυτό που ισχύει για την ιατρική, το ίδιο ισχύει και για την ε, τοξικολογία. Χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο εναλλακτικέ μεθόδου για να εξετάζουμε τα αποτελέσματα μια νέα χημική ε, ουσία. Ε, όχι μόνο πειράματα in vitro, αλλά όλο και περισσότερο προσωμιώσει με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτέ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην τοξικολογία και επίση για να εξεταστούν πιθανέ αντιδράσει με άλλε χημικέ ουσίε αλλά οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα ε, μας λένε ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε ή να σταματήσουμε πλήρως ακόμα τα πειράματα σε ζώα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ε, εξετάσει και στο πλαίσιο του ε, κοινού κέντρου έρευνας που συντηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικές φορές τα αποτελέσματα στα ζώα μπορεί να είναι πολύ περιορισμένα στο τοπικό επίπεδο. Ε, κάποιος αν ελέγχουμε μια ουσία συγκεκριμένη. Αλλά εάν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μια χημική ουσία σε έναν οργανισμό, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ε, περιοριζόμενοι μόνο στι εργαστηριακέ in vitro μεθόδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα. Ε, λέτε ότι βασιζόμαστε τοξίστη 21, το οποίο, περιπτώσει για την τοξικολογία, το οποίο θέτει το πλαίσιο. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν έχουν στόχο να γίνεται μια πρώτη εξέταση των ουσιών και να μην χρειάζεται να γίνονται πειράματα σε ζώα για όλες από αυτές, αλλά να μπορούν να περιορίζονται και να γίνονται μόνο σε ορισμένες από αυτές. Γίνεται ε, μια αξιολόγηση λοιπόν κινδύνου. Ωστόσο, τα... όταν γίνονται, χρειάζεται τελικά να γίνουν πειράματα σε ζώα, οι απαιτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ παρόμοιε με εκείνε που υπάρχουν στι ΗΠΑ. Τα στοιχεία που σας έδωσα τώρα είναι εκείνα τα οποία είχαμε αναφέρει και στην πρώτη ε, αναφορά, στην απάντησή μας στην πρώτη αναφορά, γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω αλλά όσον αφορά τον REACH, τον κανονισμό REACH και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα επικυροποιεί αυτά συνέχεια την νομοθεσία με βάση τις επιστημονικές ε, πληροφορίες, ενώ οι, οι προσφεύγουσες μας παρουσιάζουν παροχημένα επιστημονικά στοιχεία, τα μοντέλα έχουν ε, ξεπεράσει αυτά που αναφέρουν οι προσφεύγουσες και θα έλεγα ότι ο ίδιος ο κανονισμός Rich είναι πολύ πιο μπροστά από αυτά που αναφέρονται στην αναφορά. Και έχει εξάλλου και ο ίδιος επικαιροποιηθεί. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η συνοπτική έκδοση. Σας ευχαριστούμε για αυτόν τον απολογισμό που κάνατε των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας και ίσως αυτό να δώσει την έμπνευση και την, ε, να, να, να ε, την επιθυμία στις προσεύγουσες να επανεξετάσουν την αναφορά τους. Ο λόγος του συναδέλφου. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ε, ε, έχω συμμετάσχει στο Συμβούλιο ε, Ηθικής Αξιολόγησης στη, στη Δανία για τα πειράματα σε ζώα και εκεί έμαθα ότι αν κάποιο στηρίσει τους κανόνες του ΟΑΣΕ για τα πειράματα στα ζώα, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, πολύ, πολύ σαφής κανόνες που διαφέρουν από αυτό που θα μας παρουσιάζετε στο βίντεο. Για παράδειγμα, απαγορεύεται να υποβάλει κανείς σε πόνο τα ζώα. Ωστόσο, μερικέ φορές υπάρχουν συγκρούσεις στο τι επιδιωκούμε να κάνουμε. Αν προσπαθούμε να ελέγξουμε την αποτελεσμότητα του ενό παυσίπονου, πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρί να προκαλέσουμε πόνο. Το πρώτο λοιπόν σημαντικό είναι η τήρηση αυτών των κανόνων. Δεύτερον, η ίδια η βιομηχανία, η χημική και η φαρμακευτική επιθυμεί την κατάργηση των ε, δοκιμών σε ζώα γιατί είναι πολύ ακριβές. Εάν κάνουμε τη σύγκριση του τι συμβαίνει στις, στις, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, εκεί δεν έχουν την αρχή της προφύλαξης. Δεν έχουμε την αντίστοιχη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την αρχή τη προφύλαξη που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερε και υψηλότερε απαιτήσει ασφαλεία. Στι ΗΠΑ θα συμβεί κάτι και απλώ μετά θα έρθουν οι δικηγόροι και θα επαιτήσουν αποζημιώσει. Ενώ εμεί πρέπει να φροντίσουμε να είναι γνωστά τα αποτελέσματα στου ζώντε οργανισμού πριν να τεθεί στην διάθεση μια ουσία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μάλλον εμεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου δεν υποστηρίζουμε τη βιομηχανία, μάλλον αντίπαλοι του είμαστε στο θέμα αυτό. Κάτι ακόμα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε στη Δανία για τους, τις ουσίες που διαταράσσουν ε, την παραγωγή ορμονών. Γίνεται ένα πείραμα. Μας λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία οι επιστήμονες και καταφέραμε να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία με πειράματα σε ζώα που μας έδειξαν πόσο επικίνδυνες ήταν αυτές οι ουσίες στοιχεία τα οποία θα ήθελα να τα αποκρύψουν, να τα βάλουν κάτω από το χαλί η χημική βιομηχανία. Και έχουμε τώρα στοιχεία που μας αποδεικνύουν πόσο δυσμενείς επιπτώσεις έχει στην γονιμότητα των ανδρών, Ίσως τώρα κάποιοι άντρες να μην τους ενδιαφέρει αυτό, δεν την πολύ καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Αλλά επίσης δείξαμε ότι πέρα από την ανδρική γονιμότητα υπάρχουν τις επιπτώσεις και στον εγκέφαλο των βρεφών, Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιο χρειάζεται να κάνει αυτά τα, αυτούς τους ελέγχους, αυτά τα πειράματα, προτιμώ να γίνουν σε ζώα παρά να τα μάθουμε από τα αποτελέσματα που θα διαπιστώνουμε στους ανθρώπους. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Συγγνώμη, λάθος. Η Ελεονόρα Εύη είχε ζητήσει το λόγο. Πρέπει να περιμένετε δύο λεπτά. Ελεονόρα, παρακαλώ, έχει το λόγο. Να πω και εγώ κάτι. Απόλυτα υποστηρίζω την αναφορά αυτή. Σας ευχαριστώ γιατί θίξατε το σχετικό θέμα. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ κατά την άποψή μου. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε και μια πρωτοβολία Ευρωπαίων πολιτών για τα πειραματόζωα και θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και τους επόμενους μήνες σίγουρα παρά τις διαβεβαιώσεις που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται να προσέξουμε, να προσέξουμε να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό ΡΙΤΣ που επιτρέπει παρόμοιες πρακτικές ε, πειράματα πάνω σε ζώα. Υπάρχουν, ε, γνωρίζουμε πολύ καλά, πολύ αποτελεσματικότερες εναλλακτικές μεθόδους από ό,τι σε ζώα. Αλλά δυστυχώς ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν πέρασαν από δοκιμές εκτίμησης, ενώ υπάρχουν ε, κοινοτόμες μέθοδοι, μπορούν να κάνουμε κάτι διαφορετικό από επιστημονικής πλευράς και ε, να είναι αποτελεσματικότερα από ό,τι για τα ζώα. Υπάρχουν πάρα, πολλά, πάρα πολλές χημικές ουσίες και φάρμακα κλπ που από την αρχή πάνε μέχρι την εμπορία και μιλάνε για το 0,04% φαρμάκων τα οποία συμπληρώνουν αυτή την πορεία. Εντάξει. Και θα πρέπει να δούμε ε, είναι βάρβαρη και απαρχαιωμένη αυτή η μέθοδος ε, και αντιπαραγωγική και θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. πέρα βέβαια από τα πειράματα σε ζώα από ηθικής πλευράς είναι βάρβαρη μέθοδος. Πρόκειται όμως και μια πρόοδο επιστημονική για την προστασία της υγείας μας. Πέτερ, έχεις το λόγο, παρακαλώ. Ε, το μικρόφωνο του μιλητή, παρακαλώ. Πρώτη παρασύρση όταν συζητούμε αναφορά εδώ στην Επιτροπή Αναφορών, αποτελεί και μια αναγνώριση από την πλευρά των μελών ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα πρέπει κανείς να εξετάσει και από πολιτική άποψη. Αλλιώς ε, θα την είχαμε κλείσει πολύ σύντομα αυτήν την αναφορά. Επίσης, το είπε και η Κομισιόν, υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα και έχουν ε, γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν προσπάθειες να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες ε, στη βάση της μοριακής βιολογίας ενώ εξετάζεται και από πολιτικής άποψης το θέμα πώς θα μπορούσαμε αν όχι να απαγορεύσουμε τουλάχιστον να περιορίσουμε τα πειράματα σε ζώο και είπε και η Κομισιόν ότι βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εξέτησης και επικαιροποίησης της νομικής βάσης για τον κανονισμό REACH και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τον, την συμβαστική λύση. Αφού δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, να εξαλείψουμε πλήρως τα πειράματα στα ζώα, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να τα περιορίσουμε, να μην γίνονται επαναληπτικές δοκιμές σε περιπτώσεις πολλές, όταν έχει, να μην επαναλαμβάνονται πειράματα σε ζώα τακτικά ή θα μπορούσαν ας πούμε να γίνονται τα πειράματα σε ζώα όχι παντού στην Ευρώπη αλλά σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θα οριστεί στην Ευρώπη και θα μπορούσαν βεβαίως να ε, μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της ε, σύγχρονης τεχνολογίας. Αν δηλαδή διαπιστωθεί ήδη στο επίπεδο το μοριακό ότι κάποια χημική ουσία είναι επιβλαβής, τότε δεν θα χρειάζεται, να μην χρειάζεται να γίνεται και πείραμα σε ζώο. Κάνουμε δηλαδή από τη δική μας πλευρά αυτό που μπορούμε. Εμείς προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και να λάβουμε υπόψη μας μάλλον τις δικές σας ανησυχίες και τους προβληματισμούς που μας εκφράσατε και ε, πιστεύουμε ότι με αυτό το πνεύμα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πρόκειται για πραγματικά σοβαρότατο θέμα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορούμε να παραπέμψουμε τους ε, αναφέροντες και στο εξής στις 11 Μαΐου θα γίνει μια δημόσια ακρόαση που μάλιστα θα μεταδοθεί και μέσω διαδικτύου για το δικαίωμα υποβολής αναφορών με τίτλο Vivisection. Ακούσαμε λοιπόν τη δική σας άποψη, ακούσαμε την άποψη της Κομισιόν, υπήρξε δυνατότητα να γίνει συζήτηση εδώ μεταξύ των Ευρωβουλευτών και σας διαβεβαιώ ότι η δική μας η Επιτροπή θα... Ε, συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν την δημόσια ακρόαση το Stop Section οπότε θα έλεγα να τελειώσουμε τη συζήτηση ε, για τώρα και θα το επανεξετάσουμε το ζήτημα σε επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ε, εύχομαι να έχετε ένα καλό ταξίδι επιστροφής. Ελπίζω να συνεχίσετε το έργο που έχετε ήδη αναλάβει και ελπίζω να δείτε και λίγο τις Βρυξέλλες μιας και ήρθατε εδώ. Λοιπόν, επί, επόμενη αναφορά, ο κύριος Ερνέστο Σόχο είναι εδώ για την 0508 του 14 σχετικά με τη διαφθορά και, την, ε, και ε, τις εγκληματικές ενέργειες στην ε, Ρουμανία. Συγγνώμη, μπορώ να σας διακόψω. Ε, τι θα γίνει, ποια, ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί στη δική μας αναφορά. Ναι, λέει η Πρόεδρος. Σας ακούσαμε, ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι θα μεταφέρουν τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα στην ακρόαση που θα γίνει. Οπότε η αναφορά που υποβάλατε εσείς θα μας χρησιμεύσει στη συνέχεια που θα δοθεί στον, στον, στην συζήτηση αυτή. Ε, και δίνω το λόγο τώρα στον επόμενο αναφέροντά μας, τον κύριο Σόχο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Σόχο λόγω της υγείας του επειδή υποφέρει από προβλήματα ε, έχασε τα υπάρχοντά του πραγματικά στη Ρουμανία ε, μάλιστα με συμμετοχή, με συνεργασία δικαστικών αρχών και αστυνομικών αρχών. Έχει καταστραφεί ο κύριος Σόχο, έχει χάσει 2 εκατομμύρια ευρώ, ήταν αυτά που είχε επενδύσει στη Ρουμανία. Δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου, γι' αυτό ακριβώς σας πω πολύ σύντομα τα πράγματα. Τα κύρια ε, σε 11 τουλάχιστον δικαστικές διαδικασίες συμμετείχε, αλλά δεν τον καλούσαν καθόλου και το 2000 προχώρησε στη σύσταση μιας κορδέλας κοπής και επεξεργασίας μετά ξύλων σε μια από τις πιο μειονεκτικές περιοχές, την Κάρα Σεβερίν. Αλλά ήδη από το εμπορικό μελτίο της Ρουμανίας τον κορόιδεψε ο νομικός εκπρόσωπος και από την διοίκηση λοιπόν ε, του έτρωγαν σε εισαγωγικά τα χρήματα από διοικητικούς παράγοντες κλπ. Το 2002 μετά από δύο χρόνια που κατάλαβε τι γινόταν πήγε στα δικαστήρια αλλά παρόλα αυτά συνεχίστηκαν αυτές οι ανομαλίες. που τον καλούσαν με ψευδή έγγραφα ε, είτε με παρουσία ατόμων που δεν τον εκπροσωπούσα πραγματικά, δεν τον εκείνοναν τα αποτελέσματα, τίποτα, τις αποφάσεις. Ο κύριος ε, Σόχο ε, κατέθεσε και έγγραφα από το δικαστήριο της Χαγής. Του είπαν όχι είχαν πει τότε ότι α, δεν έγινε, αυτό έγινε εκπρόθεσμα. Έτσι ο κύριος Σόχο σε πολλές ε, δίκες δεν παρέστη καθόλου, δεν τον καλούσαν και ο ίδιος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του είπε «Α, δεν θα κερδίσεις γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν δώσει 24.000 ευρώ στις δικαστικές αρχές για να βγάλουν αρνητική απόφαση». Πολλές φορές λοιπόν δεν ήταν παρόν, δεν ήταν παρόν που ούτε μάθαινε καθόλου τις αποφάσεις. Και για 4.000 ευρώ που τον έκλεψαν έκανε μία μήνυση και έκρυψε τη μήνυσή του η αστυνομία και μετά υπέγραψαν ε, δήθεν ε, εκ μέρους του κλπ. και το έκρυψαν και μετά τιμώρησαν τον αστυνομικό που το ε, έκρυψε αυτή τη μήνυση. Και ο κύριος Σόχο ήρθε σε επαφή αλλά και ήδη έχουν ε, τιμωρηθεί και αστυνομικοί για όσα του έκαναν, για όσα του προκάλεσαν. Ε, υπήρχε και συνεργασία στην απάτη από έναν δικαστή και μάλιστα ένας άλλος δικαστής έκανε μια ψεύτικη δήλωση κλπ. και παρανόμως συμμετείχε στην ε, σύνθεση του δικαστηρίου και άλλοι δύο τιμωρήθηκαν για διαφθορά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν ε, σοβαρές αφιβολίες όσον αφορά τη σοβαρότητα της διαδικασίας. Πολλές φορές ε, δεν υπάρχουν και τα πρακτικά και οι διοικητικές πράξεις δεν ε, δημοσιευόταν. Όσε ήταν μόνο υπέρ των αντιπόλων του. Και δεν υπάρχει ε, κανένα στοιχείο πολλές φορές ε, και επίσης συστηματικά τον παρεμπόδιζαν να παρουσιαστεί στη δικαιοσύνη χάρη στη συνεργασία προσωπικού από την αστυνομία, από τις δικαστικές αρχές. Χωρίς να μια τέτοια συνεργασία δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν. Όλα αυτά τα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακριβώς στα πλαίσια έκθεσης της για την διαφθορά στη Ρουμανία αυτά τα χρόνια και το 2004 στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού Αντρίον Ναστάσε ε, υπέβαλε μια αναφορά, ο οποίος καταδικάστηκε Αντρίον Ναστάσε τελικά για διαφθορά αλλά τον παρεμπόδιζαν. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην διαδικασία προένταξης υπήρχαν τρεις διαφορετικές οργανισμοί για να ελέγχουν τη διαφθορά. Εκεί προσέφυγε ο κύριος Σόχο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε δώσει αρκετά χρήματα για τη μάχη κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία και η πρεσβεία της Ισπανίας παρουσίασε στον ε, Γενικό Εισαγγελέα την έκθεση σχετικά με τα γεγονότα αυτά και μετά όμως είπε ότι δεν ήταν δική του αρμοδιότητα. Μετά πήγε στη Δημισοάρα και μετά του είπαν ότι εντάξει υπήρξαν κάτι δίκες αλλά τίποτα περισσότερο δεν του είπαν. Και ο πρόξενος με συναντήθηκε με τον Γενικό Εισαγγελέα, ενημέρωσε τον κ. Σόχο ότι δεν θα γίνει τίποτα και επίσης ο μόνιμο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή στη Ρουμανία είπε ε, ο κύριος Τζόναθαν Σίλιν είπε στον κύριο Σόχο ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καμία δεσμοτά δηλαδή να καταδικάσει, να καταγγείλει αυτή τη διαφθορά. Όλα αυτά ήταν γνωστά από τότε ότι συνέβαιναν στη Ρουμανία. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί ο κύριος Σόχο τον εαυτό του και τα άρθρα 20 και 47 του Ευρωπαϊκού Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν γίνονται σεβαστά ακριβώς ζητάει ο κύριος Σόχο να ξεκινήσει μία ανάκριση ανεξάρτητη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα για να δούμε τις παραλήψεις ε, του Ρουμανικού κράτους και επίσης ζητάει μια ενημέρωση τι μπορεί να κάνει ένας Ευρωπαίος πολίτης ε, όταν ε, υπάρχουν παρόμοιες ενέργειες καταδικαστικές για τις υποθέσεις του σε ένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παραβίαση των συνθηκών. Ο κ. Γκαρσία τον κύριο Γκαρσία τον ευχαριστούμε εκ μέρους του κύριου Σόχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Κύριος Γέγκερ. Κυρία Γέγκερ, συγγνώμη. Καλημέρα σας. Με ακούτε, με ακούτε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την αναφορά αυτή. Λυπάμαι, λυπάμαι από όλα αυτά που έχετε υποστεί για τα χρήματα που χάσατε. Αλλά το είπαμε ήδη στην γραπτή της απάντησης στην Επιτροπή. Δεν είναι αρμόδια Επιτροπή. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε παρόμοιες ε, ε, προσφυγές που δεν έχουν σχέση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια προσφυγή κατά του Ρουμανικού κράτους για αυτό το θέμα. Αλλά όμως μας έχει βεθτοποιηθεί το θέμα σας όπως και άλλες παρομές περιπτώσεις που μας αναφέρονται συχνά, συνεχώς μπορώ να πω. Και λέτε η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ένα έλεγχο όσον αφορά διαφθορά στη Ρουμανία. Εάν το κάνουμε, ναι, κάνουμε αυτόν τον έλεγχο τακτικό έλεγχο για τη δικαστική εξουσία, όλα αυτά μέσω μηχανισμών συνεργασίας ε, επαλήθευσης στο CVM και ακριβώς το 2007 στην ένταξη της Ρουμανίας ε, εγγενιάστηκε αυτό ώστε να μπορέσει να δώσει τη μάχη της Ρουμανία κατά της διαφθοράς ε, το CVM κάνει μια εκτίμηση της πρόοδου που επετέχθη και μέσω μια σειράς benchmark και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ανήκω και εγώ αρκετές φορές επισκέπτονται ετησίως τη Ρουμανία και μάλιστα με εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη-μέλη και αυτό για να δούμε πώς έχει προοδεύσει η κατάσταση σε σχέση με αυτές τις νομικές μεταρρυθμίσεις και τη μάχη κατά Και ετησίως υιοθετούμε από την Επιτροπή μια έκθεση με συστάσεις προς τη Ρουμανία. Η τον Ιανουάριο του 2015 έχουμε τελευταία έκθεση από τη CVM πριν από μερικούς μήνες και το τελειώνει με το κάτι το σημαντικό για σας. Η πρόοδος του 2013 σε ορισμένους τομείς ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο το 2014. Άρα λοιπόν υπάρχει μια θετική τάση η οποία στηρίχτηκε με μια καλύτερη, μεγαλύτερη προσπάθεια των δικαστικών αρχών και με μια εντυπωσιακή μάχη κατά σε υψηλά επίπεδα διαφθοράς. Βέβαια χρειάζεται περισσότερα μέτρα, περισσότερη προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Γνωρίζουμε την ανάγκη της μάχης κατά της διαφθοράς, αλλά είναι τόσο το μέγεθος του προβλήματος που χρειάζεται μια πιο συστηματική παρακολούθηση. Ναι, επετεύχθη αρκετή πρόοδος. Εδώ λοιπόν επετεύχθη πρόεδρος και περίπου 800 άτομα συνελήφθησαν ε, στη Ρουμανία για διαφθορά μαζί και με υπουργούς, με βουλευτές, με δικαστές. Περίπου 25 δικαστές καταδικάστηκαν για διαφθορά. Επετεύχθη πρόοδος αλλά είναι μακρύς ο δρόμος. Η Επιτροπή παρακολουθεί πάντα, βοηθάει πάντα τη Ρουμανία στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, εκτός από ψηβέμε, η Επιτροπή στα πλαίσια ενός συντονισμού οικονομικής πολιτικής του εξαμήνου αυτού του ε, υποβλήθηκαν συστάσεις στη Ρουμανία για τη βελτίωση του δικαστικού της συστήματος και για μάχη κατά της διαφθοράς, το είπατε πολύ σωστά, ουσιαστικά αναχαιτίζει την οικονομική πρόοδο της Ρουμανίας το φαινόμενο αυτό. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι επιτυχάνεται κάποια πρόοδος. Επίσης μιλάτε για κάτι ακόμα στην αφορά σας σχετικά με τον οικονομικό μηχανισμό Σίγουρα στον δημοσιονομικό κανονισμό και στα διαφορετικά ταμεία υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, εσωτερικές εξωτερικές διαδικασίες ε, και βλέπουμε, ανακαλύπτουμε συνεχώς προβλήματα, διαφθορά, ε, αρνητική εφαρμογή και τότε καμιά φορά διακόπτουμε τη χρηματοδότηση, την αλλάζουμε, αυτό συμβαίνει συχνά. Αυτά ήθελα να σας πω σχετικά με αυτό. Très bien, je vous remercie. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος και εγώ. Και τώρα, και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η Λίσσα Σκούνμπιλμπα έχει πρώτη τον λόγο. Muchas gracias. Ευχαριστώ και εγώ τον Νέστο Σόχο και τους ε, όσους το συνοδεύουν ε, καλώς ήρθατε απαιτώ περισσότερη αποφασιστικότητα με έλεγχο γοργό γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι ένα άτομο ε, περιπέζονται τα βασικά του θεμελιώδη δικαιώματα και όλων των Ευρωπαίων. Αυτό που ακούσαμε την Επιτροπή. Πολύ σωστά, πολύ ωραία, γενικό πρόγραμμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε όλοι μας. Δεν προσφέρει όμως απάντηση σε αυτό που υποφέρει ένας Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό που μας ζητάει εδώ στην Επιτροπή μας από ένας εύπορος επιχειρηματίας με διαθέσει και να κάνει μια δουλειά σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι στις κοινωνικές υπηρεσίες πια να το βοηθήσουν, έχει καταστραφεί και εδώ δεν είναι οι συνθήκες της αγοράς, δεν είναι η κακοδιαχείριση. Άλλωστε αυτό πρέπει να τίθεται, αυτό πρέπει να θίγεται κάθε πρόβλημα. Όπως αυτό που λέμε τώρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς η Ρουμανία είναι στο κόκκινο στην Επιτροπή Ακριβώ ακριβώς όργανος ε, το What's Human Rights ε, και βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά και στα υψηλά επίπεδα δικαστικών αρχών. Ε, χρειάζεται, έχει απαιτηθεί ενός ανεξάρτητου ιδρύματος το οποίο να προχωράει σε ένα έλεγχο, να βλέπει όλα αυτά, αν πώς μπορούν να συνδυαστούν, τι γίνεται μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας κλπ. Και, και μια καλύτερη πιο αποτελεσματική μάχη εναντίον της διαφθοράς. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις του 2012 και το 2015 του Ενωρίου. Βλέπουμε αυτά βέβαια που γίνονται. Δεν επαρκούν όμως. Βλέπουμε ότι έχει καταστραφεί ο κύριος Σόχο οικονομικά. Όλα αυτά έχουν σχέση με το πρόβλημα αυτό της διαφθοράς πάνω από 10 χρόνια πριν και η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη τότε. Ελπίζω, περιμένω σήμερα από την Επιτροπή να αναλάβει να κάνει προβεί σε ενέργειες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση για να αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για να δοθεί το παράδειγμα ακριβώ και σε άλλες χιλιάδες άτομα που δεν έφτασαν μέχρι εδώ την Επιτροπή μας και για την Πρόεδρο της Επιτροπής ε, η μόνιμη εκπρόσωπος της Ρουμανίας που λέει ότι α, δεν υπάρχουν ενδείξεις επαρκής για να μπορέσει να γίνει μια έρευνα σχετικά με αυτές τις πτυχές για τη διαφθορά στην περίπτωση του κύριου Σόχο. Θα ήθελα να πω στα μέλη εδώ της Επιτροπής μας, ο κύριος Σόχο ήρθε με όλο το φάκελό του, με όλα τα στοιχεία. Βλέπουμε ακριβώς ότι υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, κάθε ένα ξεχωριστά, κάθε βήμα που έκανε, κάθε ενέργειά του. Αυτό που σε πέντε λεπτά μέσα μας τα είπε ο συνηγορός του. Αυτή ε, μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας, να θελοτυφλούμε. Είναι μια μόνο περίπτωση, αλλά η κορυφή μιας πυραμίδας τόσων περιπτώσεων στην Ευρώπη που υποφέρουν. Δεν γίνεται έτσι με γενικά, με γενικές διαπιστώσεις. Θέλουμε μια συγκεκριμένη ακριβώς ε, γνώμη για την περίπτωση του κυρίου Σόχο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριος Ιτουγκάης. Θα έχετε το λόγο. Προσπαθήστε να μην μακρηγορήσετε για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν αλλάζουν τα πράγματα στην Επιτροπή Αναφόρων. Για δέκα χρόνια ήμουν μέλος εδώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω ακριβώς το προσωπικό, τους συναδέλφους, παλιούς συναδέλφους κλπ. της Επιτροπής Είδαμε το τι γινόταν εδώ επί χρόνια με πάρα πολλές αναφορές και κυρία Πρόεδρε έχουμε εδώ μια αναφορά ενός Ισπανού πολίτη. Επιτρέψτε να σας πω ότι αποτελεί μια προσωπική τραγωδία για εκείνον, οικονομική τραγωδία και επιχειρηματική τραγωδία βλέπουμε τη διάλυση ενός συστήματος, την κακή λειτουργία του που κανονικά έπρεπε να είναι δημοκρατικό, δίκαιο μιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρουμανίας και για οποιοδήποτε άλλο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως το είπε πολύ σωστά η κυρία η συναδελφός μου, η Ισπανίδα, εδώ, με αυτά τα στοιχεία ήρθε εδώ, με όλα το φακελό του για να δείξει αυτή την αντιμετώπιση του ότι ε, καταπατήθηκαν τα δικαιώματά του τα δημοκρατικά. Και κύρια Πρόεδρε, ο κύριος ε, Σόχο είναι, ο παθών, αλλά αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε επιχειρηματίας, οποιοδήποτε πολίτης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή στη Ρουμανία. Επιτρέψτε μου εν συντομία κύριε Πρόεδρε να απαντήσω κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού την άκουσα πρώτα βέβαια ότι εδώ σημαίνεται μια αντίφαση εδώ της Επιτροπής της όταν μας λέει αυτά τα πράγματα ότι δεν είναι αρμόδια για να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία ναι αλλά εδώ μια και να το πω και λατινικά, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Εδώ πρέπει να δούμε. Για να εδώ στην Επιτροπή Αναφορών μας εξηγούν, ναι εντάξει, στη Ρουμανία είναι, γίνεται μια κάποια έρευνα, δεν ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, θα παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επισκέψεις σας στη Ρουμανία θα πρέπει να συμπεριλάβετε και αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση αναφορά. Αυτά που λέει ο κύριος Σόχο εδώ δημόσια, εδώ μπροστά στην Επιτροπή μας Αναφορών. Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Θα ήθελα να ζητήσω πολλά και διάφορα από την Επιτροπή Αναφορών σας. Να παραμείνει ανοιχτή η έκθεση, η αναφορά αυτή για την οποία μιλάμε. Επίσης, ε, να ζητήσουμε από ρουμανικές αρχές να έρθουν εδώ, όπως το έκανα και αρκετές φορές πριν, όταν εγώ συμμετείχα σε αυτή την επιτροπή μέλη από τις, ε, ναι, από τις αρχές και από όπως έχει γίνει και από τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία. Υπήρξαν ε, μέλη της διοίκησης που ήρθαν εδώ και μας εξήγησαν πράγματα για παρόμοια εκτρή περίπτωση όπως αυτή εδώ. Σημαντική ταυτόχρονα θέλουμε μια ξεκάθαρη δήλωση σχετικά με όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα σαν επιχειρήματα και σαν στοιχεία και ότι δεν θα πάει τώρα, ε, ξεχαστεί. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την αναφορά. Και κύρια Πρόεδρε, να σταλεί μια επιστολή από δική σας πλευράς, επιτρέψτε μου να το προτείνω αυτό κύρια Πρόεδρε, στις ρουμανικές αρχές, ε, στις ε, ε, αρχές και στις δικαστικές αρχές της Ρουμανίας για να ζητήσουμε τι ζητάμε εδώ ότι μας ανησυχεί αυτή η περίπτωση του κυρίου Σόχο και ότι οπωσδήποτε εμείς παρα, εμείς διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά αυτή για να ξέρουμε, να μάθουμε τι γίνεται, πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, τι κατάληξη θα έχει από τις ρουμανικές αρχές. Ναι, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε έτσι να κλείσουμε την αναφορά αυτή από τη στιγμή που δεν θα έχουμε μία σχετική διευκρίνηση από πλευράς των ρουμανικών αρχών. Τι ακριβώς έχει γίνει με την περίπτωση Σόχο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ακόμη ομιλητές στον κατάλογο. Συμφωνείτε να κλείσω τον κατάλογο ομιλητών μετά. Ο κύριος Ντεμπέγα, ο κύριος Μαρτάν και ο κύριος Τεριμπράχα, Τερικάμπρας. Συμφωνείτε να κλείσω τον κατάλογο ομιλητών μετά από αυτό. Κύριε Ντεμπέγα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι για αυτά που υπέστη ο κύριος Σόχο. Η, την επιχείρηση του ξεκίνησε το 2000 και από τότε στη Ρουμανία είχαμε πολλές και διάφορες μεταρρυθμίσεις όπως μια πολύ σημαντική του δικαστικού συστήματος, το είπε μόλις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τελευταίο έκθεση περί ελέγχου, παρακολούθηση λοιπά, Υπήρξε πρόοδος, φάνηκε προς την σωστή κατεύθυνση του συστήματος αυτού. Αλλά οι αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας ε, τι έγινε, έστειλαν μία απάντηση, έστειλαν μία απάντηση αλλά χωρίς όμως συγκεκριμένα στοιχεία. και σε εθνικό επίπεδο ρουμανικό ο Σόχο μετά από όσα έχει κάνει εκείνη θα μπορούσε να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα μπορούσε να αποφανθεί σχετικά με το μη σεβασμό της σύμβασης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Αφέροντα το έκανε αυτό, προσέφυγε στο δικαστήριο αυτό και τι ακριβώς πέτυχε. Και ακόμη κάτι. Η Ρουμανία έχει οθετήσει ήδη μέτρα μέσω του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου στο εδαφός της. Η έκθεση Επιτροπής Ευρωπαϊκής λέει ότι προχωράνε θετικά τα πράγματα στη Ρουμανία. Να επαναλάβω ότι λυπάμαι πάρα πολύ για όσα υπέστη ο κύριος Στόχο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάντως ε, από οποιαδήποτε χώρα και προέρχονται οι αντιδράσεις και εξηγήσει από διάφορες χώρες. Ευχαριστώ. Ο λόγο στον κύριο Μαρτάν. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα κρίνουμε εδώ τα γεγονότα. Δεν είμαστε οι αρμόδιοι. Ακούσαμε όμω τον αναφέροντα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημαντικό στην όλη συζήτηση ποιο είναι, αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή ότι υπάρχει διαφθορά στη Ρουμανία. Έτσι, αλλά δεν απαντάει σε αυτά που ρωτάει, ζητάει ο κύριος Σόχο που λέει ότι εδώ πέρα καταπατήθηκαν τα δικαιώματά μου και η Ρουμανία δεν τα σέβεται αυτό κυρίως το να έχω μια δίκαιη κρίση, μια δίκαια ακριβώ και να υπάρχουν από δική μου πλευρά όλα τα στοιχεία που θα αποδείξουν ότι ε, ήμουν θύμα απάτης κλπ. κλπ. Να λοιπόν που ισχύουν πια αμφιβολίες. Από τη στιγμή που ισχύουν αυτές οι αμφιβολίες, οι αμφιβολίες είναι υπέρ του θύματος. Στην περίπτωση του κυρίου Σόχο, εντάξει δεν είμαι αρμόδιος εγώ για να κάνω μια εκτίμηση όλων αυτών των τεκμηρίων της ε, υπεράσπισης, αλλά εδώ Άκουσα και αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να απαιτηθεί η δυνατότητα μια ειδική έρευνα για την περίπτωση κ. Σόχο. Δεν είναι έτσι. Απαντήσαμε γενικά από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαφθορά γενικά στη Ρουμανία ότι απαντάμε έτσι σε μια συγκεκριμένη αναφορά αυτή που, κάνει, που υποβάλλει ο κ. Σόχο εδώ για συγκεκριμένα δικά του ε, θέματα. Απαντώντας του καθησυχάζουμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι ένας μόνο. Είναι μια ήπειρος όπου παντού εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και γίνονται σεβασμένα αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και θα πρέπει να δούμε ε, αν δεν μπορούμε να πετήσουμε μια νέα δίκη από τη Ρουμανία τουλάχιστον ε, να υπάρξει μια κατάλληλη σωστή έρευνα ανάκριση σχετικά με αυτά. Σας ευχαριστώ, κύριος Τέρι Κάμπρας. Μην ανησυχείτε για το όνομά μου. Ε, οι φίλοι μου με αποκαλούν Τέρι. Να πω κάτι στην Επιτροπή Ευρωπαϊκή. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Μαρτέν και φίλοι μου οι Τοργάες και οι υπόλοιποι Ισπανοί που είπαν δεν φτάνει εδώ να πούμε «Α, εντάξει, γενικά η Ρουμανία προχωράει, καλά τα πάει». Είναι ένας πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται εδώ, μας διηγείται τι έγινε και τι έγινε το 2000. Δεν έχει σημασία η χρονολογία, η ημερομηνία. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκή πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε έρευνα η ίδια. Μπορεί όμως να ζητήσει η ρουμανική κυβέρνηση να διεξάγει αυτή την έρευνα για αυτή την ειδική περίπτωση να ανταποκριθεί σε αυτό και να προσφέρει εξηγήσει στην αναφορά του κ. Σόχο. Γι' αυτό θα πρέπει η αναφορά του κ. Σόχο να παραμείνει ανοιχτή, να περιμένουμε ποιε είναι οι εξηγήσει και μετά να απαντήσουμε. Ο κ. Σόχο έχει ισχυρά επιχειρήματα που προβάλλει και η κυβέρνηση ρουμανική τι λέει, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η, Ευρωπαϊκή, η ρουμανική κυβέρνηση τι λέει πάνω σε αυτό. Αυτό θα πρέπει να το ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό να ισχύει για τους υπολείπους ε, πολίτες. Είναι εδώ μια επιτροπή αναφορών που ισχύει, που έχει αρμοδιότητα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Μας τελειώνει ο χρόνος. Έκλεισα τον κατάλογο μιλών πριν από λίγα λεπτά. Οπότε δίνω τώρα το λόγο και πάλι σε εσά ως ε, δικηγόρο του κυρίου Σόχ. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω. Η Ευρωπαϊκή Τροπή που πρέπει να υπερασπίζεται τις συνθήκες, τι κάνει. υπερασπίζεται το κράτος μόνο και όχι τους πολίτες που λέει ε, δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Εδώ είναι γραφειοκρατική πολιτική η ιδέα αυτή. Αλλά σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 47 που είναι υποχρέωσή της δεν τα σέβεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν ε, η νομικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν να συντάξουν μία έκθεση για να δουν τι γίνεται ακριβώς για την παραβίαση των άρθρων 20 και 47. Γιατί ο μόνο μόνος τρόπος για να πετύχουμε κάτι το θετικό για μία πρόσβαση στη δικαιοσύνη κάτω από τις συνθήκες αυτές. Και να ολοκληρώσω κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα να καταχρωστώ του χρόνου σας, δεν ήθελα να πω τίποτα περισσότερο, αλλά ανησυχώ, σας το λέω ειλικρινά, ανησυχώ για αυτά τα Ρουμανίας. Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ακριβώς ότι όταν υποβάλλουμε στη Ρουμανία διάφορα επίσημα έγγραφα εξαφανίζονται και αυτό δεν βοηθάει στην έρευνα την όλη. Έχει γίνει αυτό, έχουν εξαφανιστεί έγγραφα. Συνάδελφοι, ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ευαίσθητο λεπτό ζήτημα. Οπότε θα ήθελα να με ακούσετε παρακαλώ για να μεταφέρετε και το μήνυμά μου στον πελάτη σας. Ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ λεπτό και πολύ δύσκολο ζήτημα. Και πραγματικά συμπάσχουμε με τον κύριο Σόχο που έχει πληγεί σημαντικότατα. Θα προτείναμε η Επιτροπή μας να δώσει εντολή στην Γραμματεία να συζητήσει με την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου ενδεχομένως να βρεθεί ένας τρόπος για να δοθεί συνέχεια στο ζήτημα, ταυτόχρονα να διατηρηθεί ανοιχτή η ε, αναφορά σας. Ίσως θα μπορούσαμε να αποστείλουμε μια επιστολή εκ μέρους της Επιτροπής μας στον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά θα ήθελα πρώτα να δούμε τι θα, σε ποια αποτελέσματα θα καταλήξουμε μέσα από τη συζήτησή μας με την νομική υπηρεσία. Θα μπορούσαμε επίσης να αποστείλουμε επιστολή στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρουμανίας και να ζητήσουμε οι αρμόδιες αρχές να τοποθετηθούν για αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό μπορώ εγώ να προτείνω ως συνέχεια. Βλέπω ότι ενδεχομένως δεν σας ικανοποιώ, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Οπότε, εντάξει, αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη στην σε διάταξη. Καλό ταξίδι, επιστροφή στην Ισπανία. Και σας παρακαλώ να μεταφέρετε από τη δική μας πλευρά τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Σόχο, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και των ε, Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ και πάμε στην στο επόμενο θέμα, στο 12 Έχουμε συζητήσει ήδη τη γνωμοδότηση για τη συνέχεια που εδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το δικαίωμα στο νερό. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν χρειάζεται να γίνει επί τη ουσία συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται να διευκρινιστεί είναι ότι η επόμενη η διαδικασία στο εξή θα είναι εξή. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση θα γίνει εδώ στην Επιτροπή στις 5 Μαΐου και ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε μια εξαιρετική γνωμοδότηση. Να πω ένα πράγμα μόνο. Έχω ήδη μία, έχουμε ήδη κάνει μία προκαταρκτική συνάντηση με τους σκιώδους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ναγκής. Δεν είναι εδώ, αλλά μου έστειλε μια εξαιρετική επιστολή, την έλαβα σήμερα το πρωί ή χθες, δεν θυμάμαι. Και απλά θα ήθελα να πω ότι περιείχε πραγματικά πολύ επικοδομητικές σχέσεις. Θα ανυπομονώ να δω τις τροπολογίες και προγραμματίζεται συνεδρία συνάντηση των συντονιστών των σκιωδών, με συγχωρείτε, την επόμενη εβδομάδα και για το ζήτημα του κανονισμού για τις ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες πολιτών ε, θα σας μιλήσει ο συνάδελφος. Οπότε, ωραία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Πάμε στην επόμενη γνωμοδότηση. Πέτερ, γρήγορα. Ο, ο, ο συνάδελφος Νάτζη είναι άρρωστος, γι' αυτό λείπει. Αυτό ήθελα απλά να διευκρινίσω. Okay. Εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι η συνεργασία θα είναι εξαιρετική. Και τώρα για την πρωτοβουλία πολιτών Ελπίζω να, να, να το προφέρω σωστά το όνομά της. Είναι η ε, γνωμοδότηση και ε, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 23 Απριλίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, αναφορών θα γίνει στις 23 Ιουνίου, ενώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων η ψηφοφορία θα γίνει 22 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι, απλά ήθελα να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα. Και με αυτό με χαρά κηρύσω τη λήξη της συνεδρίασης, της πρωινής συνεδρίασης. Θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα με τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.